Υπάρχουν κάποιοι που είναι όλη μέρα εδώ και θέλουν να τελειώσουμε στην ώρα μας. Θα είμαι κι εγώ αυστηρός λοιπόν. Υπάρχει μια ανακοίνωση πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης από τις ομάδες ε, ΕΛΚ, Σοσιαλιστών, ECR, ε, λάβα ε, στοιχεία σχετικά με διορισμούς θα δημοσιευτούν και αν μέχρι την έγκριση των πρακτικών δεν υπάρξουν ενστάσεις, οι διορισμοί θα ισχύουν ως εγκεκριμένοι. Προχωρούμε. Προφορική